απαλλαγή για το 2017 είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, ξεκάθαρα να ενισχυθεί και να είναι πιο αποτελεσματικός παγκόσμιος παίκτη. από πλευράς ε, ασφαλείας αλλά και ως μεγαλύτερος χορηγός θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις, ε, τα προγράμματα χρηματοδότησης με χώρες εταίρους. Ιδάλλως θα δώσουμε μια εικόνα ότι κάπως φυτρώνουν στα δέντρα τα χρήματά μα, ενώ αυτό δεν ισχύει. Το ερώτημά μου προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τι ε, δαπάνε αυτέ. Πώ θα αντιμετωπίσετε την έλλειψη προβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιο χρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα, Θα κάνετε μία εκτενή και ε, εκβάθρον αξιολόγηση προκειμένου να έχουμε μία προσέγγιση βάση των επιδόσεων. Μετά τώρα, από μία επιστολή που έλαβα από την ύπατη εκπρόσωπο, θα μπορούσατε να μου δώσετε μία ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ό,τι αφορά τους παρόχους υπηρεσιών για τις ε, αποστολές εκλογικών παρατηρητών. Ο κύριος Δέβα δεν είναι εδώ. Λεοντίνη από την Επιτροπή Μεταφορών. Για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έχει το αποκλειστικό νόμιο να εγκρίνει την εκτέλεση του προπολογισμού ω ένα θεσμικό όργανο άμεσα εκλεγμένο από του πολίτε, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο έτσι ώστε να εγγυηθεί ότι τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζονται σωστά τα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία απαλλαγή για το 2017, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλιση Αεροπορία, ε, για του σιδηρόδρομου, ε, τη της κοινή επιχείρησης ΣΕΖΑΡ και το ΣΥΠ του ΡΕΙΛ βασίστηκα στις αιτήσεις έκθεσης του Ευρωπαϊκού Λεκτικού Συνεδρίου. Διαπίστωσε ότι οι δύο κοινέ επιχειρήσεις και οι δύο οργανισμοί έχουν διαχειριστεί τον προπολογισμό τους με νομιμότητα. Έτσι λοιπόν πρότεινα την απαλλαγή καλώντας αυτούς τους οργανισμούς να συνεχίσουν στην ε, οδό της διαφάνεια διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ευχαριστώ. Για την Επιτροπή Ρέτζη, κυρία Μιχαηλόβα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Συνεδρίου, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης με τα τονίζει την μείωση του ποσοστού σφάλματος σε ό,τι αφορά την εδαφική συνεργασία και συνοχή μάλλον. Είναι πολύ σημαντική η μείωση. Από το 4,8 πήγαμε στο 3% για το 2017. Όλα αυτά τα σφάλματα σε επιλέξιμες δαπάνες συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στο συνολικό υπολογισμό του σφάλματος. Έχουν ληφθεί πολλά μέτρα για τον μετριασμό των συνεπειών των σφαλμάτων. Και εν και της ενδιάμεσης ε, αναθεώρησης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου ε, ε, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, αλλά χρειάζονται και άλλα και περισσότερη ευελιξία. Ευχαριστώ η κυρία Πετήρ, εξ της Άγκρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο τρόπος που διενεργούμε αυτές τις απαλλαγές παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις προς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται με διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η καλύτερη ταυτοποίηση των αιτιών των σφαλμάτων είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει το Ενεκτικό συνέδριο να ελέγξει γιατί προέκυψαν τα σφάλματα. Έχουμε σύνθετες διαδικασίες με πολλούς συμμετέχοντε. Ε, εκεί λοιπόν είναι αρκετά πιθανό να υπάρχουν ε, κατά λάθο τέτοια σφάλματα. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα περιθώριο απάτη σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Η κοινή γεωργική πολιτική επηρεάζει 11 εκατομμύρια γεωργού, παραγωγού και 22 εκατομμύρια υπαλλήλου στο γεωργικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τα σφάλματα να εντοπίζονται εν γέρος. Ευχαριστώ κύριο Καντέκ από την Επιτροπή Αλία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Αιλία κάθε χρόνο γνωμοδότησε σχετικά με την απαλλαγή για την γενικό προπολογισμό τη Ένωση. Φέτο η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά το έτο 2017 δεν ε, ε ιδιαίτερης ε, ιδιαίτερων σχολείων. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή Αιλία θα ήθελε να παρουσιάσει το Ελεκτικό Συνέδριο ξεχωριστά ποσοστό λάθο για την αλία και σε σχέση ε, και να μην είναι αυτό σωρευμένο γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια σωστότερη αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης. Η Επιτροπή Αλίας ε, θέλει να υπενθυμίσει ότι ε, η έλλειψη κατανόηση από την πλευρά του, κράτου, του κράτους μέλους, η έλλειψη συγγνώμη, ε, υλοποίηση των κονδυλίων είναι ενσχετική. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες, πάλι από την Επιτροπή Ελίας, για ένα λεπτό. Ε, ο οργανισμός Αλίας υποδειγματικά ε, εκτελεί τον προπολογισμό του οργανισμός ε, είναι σημαντικός για να καλύπτει όλο ένα και περισσότερες ευθύνες και να ρυθμίζει την εκτέλεση της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Είναι πολύ πλοκός ο τομέας της Αλίας και πολύ περισσότερο σήμερα. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η έξοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή της κοινή ελευτικής πολιτικής, η υποχρέωση εκφόρτωσης, ο κανονισμός τεχνικών μέτρων ή ε, οι ανάλογες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής απαιτούν από την Ευρώπη να μετατρέψει αυτή την πολιτική σε πολιτική προτεραιότητας. Είναι πολύ, ε, πολλά τα εδάφη όπως τα δικά μου, η Γαλλικία για τις οποίες είναι σημαντικές μια ισχυρή ελευτική πολιτική που να έχει τους απαραίτητους πόρους και να μην ε, αποτελεί αυτό αντάλλαγμα σε κάτι. Εγώ γι' αυτό εργάστηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι δίκαιο και απαραίτητο. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό για την Επιτροπή Πολιτισμού η κυρία Ντροσιεύσκη, ο κύριος Ντροσιεύσκη. Θα ήθελα... να επισημάνω δύο σημεία. Καταρχήν όσον αφορά τον προπολογισμό και τους διορμηνείς. Ε, όσον αφορά το πρώτο αυτό θέμα, θα ήθελα να πω ότι το Erasmus ε, Plus έχει εκτελεστεί, έχει υλοποιηθεί και ο τρόπος υλοποίησης είναι θετικός. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί το πρόγραμμα αυτό υφίσταται εδώ και 30 χρόνια και πάνω από 9 εκατομμύρια φοιτητές έχουν λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Δεύτερον, η Δημιουργική Ευρώπη εδώ έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι αρκετό το ποσοστό απορρόφησης 20-21% ε, και θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα ε, δεν αξιολογείται θετικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φραντς από τη ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριοι συνάδελφοι. Ως Συμβουλευτική Επιτροπή ε, διατυπώσαμε κάποιες συστάσεις όσον αφορά την παραγή χορήγηση των οργανισμών που με τη ΛΥΜΠΕ. Ε, βασικά ε, συνιστούμε τη χορήγηση απαλλαγή σε όλους τους οργανισμούς. Ωστόσο θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο. Είναι κρίμα ε, οι υπηρεσίες αυτές λόγω ανεπάρκειας χρημάτων να μην μπορούν να δημοσιεύσουν ε, στην ιστοσελίδα της ε, ΕΠΣΟ η Τσέπολ, η ΦΡΑ κλπ. Δεν μπορούν να αναρτήσουν την υποβολή υποψηφιότητα σε αυτές τις ιστοσελίδες λόγω λοιπόν πόρων και αυτό οδηγεί σε κάποιες ε, εξαρτήσεις και σε κάποιου κινδύνους ασφαλείας. Και τέλος θα ήθελα να σα επισημάνω ότι τα δείγματα ε, στην διενέργεια ελέγχων των προπολογισμών είναι τόσο περιορισμένα που είναι δύσκολο να οδηγηθούμε σε ένα σωστό συμπέρασμα. Ο κύριος Μπιούρκ για την, από την Επιτροπή Γυναικών. Η κυρία Μπιόρκ, ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ εξετάζουμε την ε, ποιότητα σε κάθε έγγραφο, αλλά όταν πρόκειται για ένα ζήτημα βασικής αποτυχίας των θεσμικών οργάνων, δεν ε, φτάνει μια ωραία διατύπωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ισότητα και χρειαζόμαστε κονδύλια δεν εξετάζουμε μόνο τα δικαιώματα των γυναικών από φεμινιστικής άποψης, δεν παίρνουμε αρκετά κονδύλια. Και η αξιολόγηση των επιμέρους ε, ταμείων ε, και το πώς επηρεάζουν την ισότητα δεν διεξάγεται. Δεν διενεργείται κανένα τέτοιο έλεγχο. Θέλουμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, ε, στην βία κατά των γυναικών, τα δικαιώματα των γυναικών στην ε, αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία. Όλα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν ε, στον προπολογισμό. Συνεχίζουμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Εξ ονόματος του ΕΛ και κυρία Γκρέσλα για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Συμβουλίου που ήρθε εδώ και που τοποθετήθηκε. Ε, και θα ήθελα να το καλέσω να συνεχίσουμε τις συνομιλίες ούτε ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δικασία απαλλαγής στο Συμβούλιο. Ε, Καλώ ήρθατε λοιπόν και χαιρόμαστε που είστε εδώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσά και την ομάδα στο επιτελείο σα. Γνωρίζουμε ότι η απαλλαγή την παίρνετε σοβαρά, γι' αυτό θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και θα ήθελα να σα παρακαλέσω στα σημεία τα οποία εξαγγείλατε, ιδιαίτερα την προκήρυξη διαγωνισμών για του γενικού ε, διευθυντέ, που είναι πιο σημαντικά από το θέμα του Γενικού Γραμματέα. Ε, να βρείτε μια λύση εδώ σε αυτή τη θητεία. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σύγκρουση συμφερόντων και επίσης ε, όσον αφορά το EG θα ήθελα να σας πω ότι έμαθα σήμερα για την EMJ ήταν ένας ε, οργανισμός ο οποίος είχε συσταθεί από την προηγούμενη επιτροπή. Ε, μου έκανε εντύπωση αυτή η απόφαση ε, και δυστυχώς δεν έχουμε καμία πρόσβαση ε, στα στοιχεία βάση των οποίων το δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση αυτή και θεωρώ ότι αυτή είναι μεγάλη έλλειψη διαφάνειας και θα πρέπει να τη διορθώσουμε. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα μισή λεπτό, κύριο από και δημοκράτε. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Είχαμε αξιοσημείωτη πρόοδο το 2017. Σκέφτομαι ότι ε, αυξήθηκε η προβολή της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρξαν προσπάθειες ε, για ε, να καλύψουμε τα έξοδα και επίσης τηλεργασία για τους υπαλλήλους, επίσης προστασία στους Βρετανούς υπαλλήλου του Κοινοβουλίου. Ε, και προστασία του σταζιέρου. Όμω πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Καταρχήν να επιτρέπουν στα πολιτικά κόμματα να λάβουν χρηματοδότηση από ιδιωτικέ επιχειρήσει. Δεν είναι αποδεκτό πώ, ε, παραδείγματο χάρη, ένα βουλευτή Επιτροπή Περιβάλλοντο θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα πολιτικό κόμμα που θα ε, χρηματοδοτείται το τη Μπάγκερ. Εγώ, εξ ονόματο τη ομάδα των Σοσιαλιστών, έχω καταθέσει μια τροπολογία ζητώντα την απαγόρευση τέτοιων επιδοτήσεων Ελπίζω να υποστηρίξει το σύνολο των πολιτικών ομάδων την τροπολογία 30 απόψε στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δεύτερη παρατήρηση. Ζητώ συγγνώμη, συνάδελφε. Α, συγγνώμη. Έχετε 1,5 λεπτό. Λυπάμαι. Έτσι λοιπόν υπήρξε διστακτικότητα στο να υπάρχει μια επιτροπή για την καταπολεμήση παρενόχλησης. Ε, όμως αυτό είναι εντικό εμείς με την κυρία Γιάλα Σέντερ, τους Πρεσίνους και την έχουμε καταθέσει μια σχετική τροπολογία. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου πρόεδρο. Και πάλι συγγνώμη. Ε, so, uh, next, uh, ο κύριος Τσαρνέσκι για το ECR για ένα λεπτό. Θα ήθελα να πω ότι επειδή μας πιέζει ο χρόνος, καθώς έχουμε ψηφοφορίες στις 5, δεν θα μπορέσω να δεκτώ έτοιμα για μπλε κάρτα. Έχετε το λόγο κύριε Τσαρνέσκη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, έχω την ε, αίσθηση déjà vu γιατί κάθε χρόνο στο πλαίσιο αυτής της ε, διαδικασίας ε, αναφερθόμαστε στην έλλειψη συνεργασίας με το Συμβούλιο. Είναι μια ιστορία δίχως τέλος, έχω την αίσθηση. Ε, δεν γίνεται εδώ καμία πρόοδος. Και πραγματικά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι ανήκουστο. Και θα ήθελα να πω το εξής. Ε, το, σε σχέση με το Ταμείο Μετανάστευσης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ε, θα πρέπει να γίνει μια διόρθωση όσον αφορά το ποσοστό σφαλμάτων. Θα πρέπει να γίνει διόρθωση. Η κυρία Διαμπάλοβα. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ δύο λόγια για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γελά Σέντερ για τη συνεργασία και την καλή δουλειά, αλλά και επειδή συνεχίσει να συνεισφέρει στην αλλαγή της αντίληψης ε, της απαλλαγής. Ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για το πώς εξοδεύουμε τα κονδύλια των πολιτών. Θα πρέπει να βρούμε τα λάθη και να τα διορθώσουμε και να έχουμε και προληπτικά μέτρα. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι μιλάμε για το λιγότερο του 3% των συνολικών δαπανών τη Ένωσης. Αν ξεχνάμε λοιπόν ότι το 97% των δαπανών ε, έχουν ε, δοθεί σωστά και εγκαίρως, όχι μόνο χάρη των, ε, στους πολίτες και για τις εταιρείε, αλλά εξυπηρετούνται και οι κοινοί μας στόχοι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτό να το παρουσιάσουμε ως επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες. Ήδη ως εισηγήτρια για την απαλλαγή 2014 για την Κομισιόν, εγώ προσπάθησα ε, να θεωρήσω ότι η απαλλαγή έχει νόημα στην αξιολόγηση το πώς δαπανούνται τα χρήματα των πολιτών. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να επικεντρωθούμε σε γεγονότα και συνδέσεις εντός του οικονομικού έτους και να μην το χρησιμοποιούμε αυτό ως ε, μία αναφορά για μελλοντικά γεγονότα που δεν έχουν καμία σχέση στη συζήτησή μας για τους πρασίνους, ο κύριος Στάς. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι σε ό,τι αφορά την σωστή διαχείριση των δημοσίων κονδυλίων, όποιο ζητά την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία πρέπει να κοιτάξει και τα του οίκου του. Γι' αυτό ω πράσινοι χαιρόμαστε που σε αυτέ τι εκθέσει εξετάζουμε διάφορα κανθόδη ζητήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την, ε, το διορισμό του κυρίου Σέλμαερ, ιδιαίτερα φιλογόμενη υπόθεση, ω Γενικού Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ήταν ένα ε, πραξικόπημα ουσιαστικά και μάλιστα ε, αναφέρθηκε και από επίσημα χείλη ότι ε, ξεπεράστηκαν τα όρια. Γι' αυτό καλούμε να εγκρίνουμε τις εφιστάμενε παραγράφους και τις τροπολογίες και να καταδικάσουμε ότι ο Σέλμαρ ήταν παρόν σε δύο συνεδριά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου προετοιμάζονταν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όποιος λοιπόν εξετάζει τα του οίκου του θα πρέπει να εξετάσει και την σύγκρουση συμφερόντων του Πρωθυπουργού της Τσεχία Μπαμπή και του, της κοινοπραξίας Agrofair που έχει λάβει εκατομμύρια ε, επιδοτήσεων. Κύριε Έτιγκερ, έχω δύο σαφή ερωτήματα προς εσάς, ελπίζω να με ακούτε. Πρώτον, ποια είναι η κατάσταση ό,τι αφορά την έρευνα και τους ελέγχους ε, διαφόρων γενικών διευθύνσεων σε, αυτές τις, αυτή την υπόθεση της Τσεχίας. Δεύτερον, πότε θα λάβουμε την τελική έκθεση. Τρίτον, θα υπάρξει απόφαση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τις ευρωεκλογές του 19. Τέλο, συνάδελφοι, και στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσουμε τα του οίκου μα μια σημαντική ε, επανεξέταση και αναθεώρηση του συστήματος αποζημιώσεων ιδίων ε, δαπανών πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Τα χρήματα που δεν δαπανώνται θα πρέπει να επιστρέφονται στο Κοινοβούλιο. Όλα τα, ε, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα διατηρεί ο δικαιούχο και θα πρέπει να ε, δημοσιεύεται και μια ετήσια έκθεση. Μόνο έτσι μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστούμε για την ΚΟΕ ο κύριος Δε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα σχόλια μου έχουν να κάνουν με την απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Και πάλι έχω αποβάλει πρόταση για την απίστευτη κατάσταση των εργαζομένων μέσω της Manpower. Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μου έχουν ε, ενημερώσει για τα κακό κείμενα. Εκφοβισμός, ε, πολύ σύντομα διαλύματα το μεσημέρι. Ε, είμαι μακρύς κατάλογος παραβιάσεων και όλα αυτά βέβαια με τον ελάχιστο κατώτατο βασικό μισθό που επιτρέπεται στο Βέλγιο. Πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση. Υπάρχει νέος διαγωνισμός, αλλά δεν ε, βρήκατε τίποτα τελικά μετά τις έρευνες που έγιναν. Γιατί όχι. Και μάλιστα έλαβε παράταση η σύμβαση με τη Manpower Solutions. Ποιε είναι οι προποθέσει που τίθενται ε, για τέτοιου είδου συμβάσεις. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να ε, παρέμβουμε. Και εμείς και ο Γενικός Γραμματέας. Ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος με το προσωπικό, με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται. Καμία προϋπόθεση διαφάνειας για τις δαπάνες. Και πάλι έχουμε υποβάλει πρόταση για αυτό το θέμα. Ελπίζω να το λάβει υπόψη και το Προεδρείο πριν το τέλος της θητείας να έχει επιληθεί το ζήτημα. Ευχαριστώ για δυόμιση λεπτά, εξ ονόματος του EFDD, ο κ. Μπουλόκ. Uh, Σας ευχαριστώ για να αναφερθώ στο τι πραγματικό συζητάμε, για όσους μας παρακολουθούν, συζητάμε την ε, απαλλαγή, τη διαδικασία της απαλλαγής των ευρωπαϊκών οργανισμών και θεσμικών οργάνων και πρέπει να δώσουμε πολιτική έγκριση. Ε, ε καθώς ε, είναι αυτό μία από τις λίγες ε, διαδικασίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, για να ελέγξουμε τους οργανισμούς. Ε, θέλω να αναφερθώ στο ΕΑΣΟ που έχει ένα προπολογισμό 86 εκατομμυρίων. Το ελεκτικό συνέδριο έδωσε αρνητική γνώμη για την ομιμότητα των πληρώμων του και έτσι αναφέρθηκε σε κακή διαχείριση των κονδυλίων και παραβίαση του νόμου, αν δούμε τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2020, θα αυξηθεί σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμω, ε, χτε το βράδυ στην Επιτροπή Προπολογισμών εγκρίνεται πάνω από 3 εκατομμύρια για 51 ε, ε, συμβασιούχους προκειμένου στα διάφορα κράτη-μέλη να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή κοινότητα εν ώψη των ευρωπαϊκών. Αυτή η μηχανή προπαγάνδας που χρηματοδοτείται από το κράτος με βρίσκει αντίθετο. Ε, θέλω να προστατεύσω τα χρήματα του φορολογουμένου. Αν συνεχίσει την προδοσία του Brexit, η Τερέσα Μέη, το θα πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση. Έτσι λοιπόν, αν περάσει η συμφωνία αποχώρηση, οι Βρετανοί φορολογούμενοι θα χρεωθούν 39 δισεκατομμύρια. Γι' αυτού του λόγου θα καταψηφίσω ε, την απαλλαγή αυτών των ευρωπαϊκών οργανισμών. Όλα ε, αυτά τα θέματα πολιτική ε, θα πρέπει να τα χειρίζονται οι εκλεγμένε δημοκρατικά κυβερνήσει, είτε μόνε είτε διμερό. Για την ομάδα ΙΕΝΕΦ, e ο κύριος Τσόκα, για δύο λεπτά. Όποιος οδήποτε έχει λογική και είναι οικογενειάρχης θα έβλεπε τις δαπάνες αυτής της απαλλαγής και θα αντιλαμβανόταν ότι υπάρχουν πάρα πολλές σπατάλες. Σπατάλες και δεν θα αρκούσε καν ολομέλεια για να τα φυγηθούμε όλα. Θα περιοριστώ σε κάποια για να σας τα υπενθυμίσω και να ελπίσω ότι κάποια λογική θα μπει στο κεφάλι όσων διαχειρίζονται αυτούς τους οργανισμούς και να μειωθούν οι σπατάλες. Ε, ε, για 48 μέρες ε, το χρόνο που χρησιμοποιούμε την έδρα του Στρασβούργου στοιχίζει σχεδόν ένα, συγγνώμη, ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε 5 χρόνια, 250 εκατομμύρια το έτος και μετακινούμαστε μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξέλλες και έχουμε 15.000 τόνους εκπομπών. Θέλει Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει το 2030 στη μείωση του 40% της ρήπανσης, εμείς δεν συνεισφέρουμε. Κατόπιν έχουμε 9 εκατομμύρια για τον οίκο ιστορίας της Ευρώπης, 200 άτομα, 9 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια για την παλιά έδρα του ΕΟΦ, γιατί ε, κάποιος ξέχασε να προβλέψει τη ρήτρα ε, της επιστροφής, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ρήτρα, θα είναι καινή θέση μέχρι το 2019. 16 δισεκατομμύρια για διοικητικές ε, δαπάνες. Αυτό προβλέπει ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, αλλά δεν σας αρκεί. Θέλετε ακόμα να ξοδέψετε 33 εκατομμύρια ευρώ για την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές σκέφτεστε να κρύψετε τις δαπάνες αυτές. Όμως είναι σαφές ότι ε, κάποιος ε, σκέφτηκε ότι δεν αντιδρούν οι λαοί. Σήμερα αντιδρούν όμως οι λαοί και είναι έτοιμοι να σας ε, καλέσουν εσάς με το κουτί της κάλπης και να σας πούνε να εγκαταλείψετε αυτό το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Τέλειωσε ο χρόνος σας. Ο κύριος Τστεχόφσκι για ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Δεν με ακούτε. Κύριε Πρόεδρε του Λεκτικού Συνεδρίου, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να υποστηρίξω την απαλλαγή για όλες τις κοινέ επιχειρήσεις και μπορώ να θεωρήσω την έκθεση αυτή ισορροπημένη συνεργασία είναι κλειδί στα πλαίσια των κοινών επιχειρήσεων για να προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Και η στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στείλει μια πολύ πιο ισχυρή εντολή στα κράτη-μέλη. Προκειμένου να ενδυναμώσουμε και να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και αν και βλέπω ότι δεν ακούτε. Θέλω να σας ε, θέσω μια βασική ερώτηση, το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Εμείς έχουμε μια πολύ σημαντική οδηγία που θα έπρεπε να το έχει καταπολεμήσει αυτό. Και ο κύριος ε, Στάς έθεσε τρεις σημαντικές ερωτήσεις σε εσά. Μόνο μία θα ρωτήσω εγώ, κύριε Πίτροπε. Αν ήδη με ακούτε. Εσείς θα καταπολεμήσετε την σύγκρουση συμφερόντων ε, κάποιων κορυφαίων πολιτικών και θα μας απαντήσετε γιατί κάποιες από τις ερωτήσεις στους πρωθυπουργούς είναι ακόμα μυστικό. Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καλό σας απόγευμα. Ε, Επίτροπε, Πρόεδρε του Ελεγκτικού, θα ήθελα καταρχήν να ε, ε σας ευχαριστήσω για τις εισηγήσει αυτές, για τις εκθέσεις. Εγώ ήμουνα από κοινού ε, συντάκτης σε μία έκθεση και τάσομαι υπέρ της ε, εσωτερικής διαχείρισης αλλά ε, περιέχονται ορισμένοι κίνδυνοι στις ε, κοινοπραξίες. Υπάρχει ένα πρόβλημα της εφαρμογής του ορίζοντα 2020, αλλά θεωρώ ότι η ποιότητα υπερέχει της ποσότητας και στόχος μας είναι να κάνουμε σωστές επενδύσεις. Όμως, το όλο εγχείρημα δείχνει την υψηλή προσθέμενη αξία αυτών των επιχειρήσεων και χαίρομαι για ότι μπορούμε να ζητήσουμε, να ζητήσουμε απαλλαγή για όλες τις εκθέσεις για το 2017. Ε, Μακοβέ. Νομίζω ότι η σύγκρουση συμφερόντων είναι ο ελέφαντας στην αίθουσα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει καμία έκθεση επί του θέματος αυτού από το 2012 όταν το ζήτησα εγώ. Άρα το ελεγκτικό ε, δεν έχει συντάξει ε, έκθεση για θέμα σύγκρουση συμφερόντων. Ε, μιλάμε για ελικόπτερα, για αεροπλάνα, για πολλαπλά προϊόντα και δυστυχώς ποτέ το ελεγκτικό δεν έχει ασχοληθεί με θέματα σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε και μία νέα μόδα τώρα τελευταία. Αυτή η ε, οργανισμοί συντάσσουν μία δήλωση έλλειψης ε, σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά αυτή είναι μία δήλωση που γίνεται τους ίδιους τους οργανισμούς. Λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να αρκείστε στο χρόνο σας. Άλλη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε Έτιγκερ, Πρόεδρε Λένε, θα ήθελα ε, να ε, ευχαριστήσω τους εισηγητές για τις απαλλαγές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους άλλους οργανισμούς. Οι οργανισμοί αυτοί βοηθούν στην καθημερινή μας ζωή έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Οι 32 οργανισμοί φτάνουν σε 2,24 δις ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες τους, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την νομιμότητα και την τακτικότητα των πληρωμών για όλους τους οργανισμούς παρά από ορισμένες αδυναμίες ως προς το προσωπικό ε, την επάνδρωση δηλαδή των οργανισμών και τις ε, δημόσιες προμήθειες βλέπουμε ότι υπάρχει μία ορατότητα. Επίσης υπήρξαν βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και προστιθέμενη αξία. Ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει θετική στάση. Φτάσαμε στους στόχους για το 2020 17 το 99% του προϋπολογισμού ε, έχει απορροφηθεί και μόνο το 1% πρέπει να ακυρωθεί. Αυτό δείχνει χρηστή διαχείριση. Και έχουμε εκπληρώσει τους στόχους προτεραιότητας. Μπορούν να γίνουν βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα του 2017, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε την ε, συνολική εργασία. Τάραντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ομάδα των Πρασίνων έχει εκφράσει κάποιε επικρίσει για την αποζημίωση γενικών εξόδων. Δεν τα επαναλάβω. Το 2017 έγινε εσωτερική ανάθεση των υπηρεσιών με τους οδηγούς και μπορεί να μην θυμάστε πόσες επικρίσεις είχαμε τότε εκφράσει όπως και εκείνη η γνώμη και ήταν κάτι που μας είχε απασχολήσει εδώ. Όμως το σύστημα αυτό στους επαγγελματίες στους οδηγούς είναι πάρα πολύ καλό. Όμως γυρίζουν άδειε οι λιμουζίνες μόνο με τον οδηγό και υπάρχουν κάποιοι που ασκούν κριτικές. Ο Βέλγος, ο κύριος Φερχόφστατ, ίσως θα μπορούσε να μάθει και στους άλλους να το χρησιμοποιούν αυτό το, το όχημα και να γυρίζουν πίσω. Θα ήθελα ε, να αναφέρω τον ε, Ρώσο Αντρέ Πλατώνοφ. Αν έχουν τα χρήματα δαπανηθεί στα χέρια της Γκουβενεό, μάλλον έχουν δαπανηθεί σωστά. Κύριος Φλάνγκαν για 1,5 λεπτό. Στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ε, ε, είμαστε ο θεματοφύλακα ε, τη εκτέλεση του προπολογισμού από την Κομισιόν και μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι δαπάνε. Η έκθεση αυτή συνοψίζει το έργο όλη τη χρονιά. Βέβαια, θα καταψηφίσω ω ηθιστέ τη χορήγηση απαλλαγή για το 2017, όμω Χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι θα πρεψηφίσω αυτήν την έκθεση που είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης δουλειά όλων των πολιτικών ομάδων, ιδίως στο έργο της κυρίας Αγιάλα Σέντερ και του προσωπικού της που κατέθεσαν μια αρχική πρόταση αλλά ακολούθησαν μια πολύ θετική προσέγγιση με τι και τι συμβιβαστικέ. Δεν είναι όλα βέβαια ρόδινα και το ελεγκτικό συνέδριο οφείλει πολλά απέναντι στους πολίτες και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσει δηλαδή τον έλεγχο ε, της Κομισιόν και των όσων δηλώνει, να είναι ειλικρινή και διαφανή. Το 2017 όμως έχουμε πάρα πολλές τρύπε και πολλά διαφανή στοιχεία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διορθώσεις ε, του περιθωρίου σφάλματος. Ε, στα 90 δευτερόλεπτα που έχω δεν μπορώ να σας πω και πολλά, απλά ότι πρέπει να εκτεθούν αυτά τα σφάλματα, όπω και πράγματι συνέβη. Ο κύριο Αλαφράγκα Σάντσερ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Αρκτικού Συνεδρίου, κύριε και κύριοι εργάστηκα για την απαλλαγή των λοιπόν οργάνων. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Νομίζω ότι οι τροπολογίες και οι λίγες τώρα στην Ολομέλεια ε, θα συμβάλλουν στη βελτίωση του έργου των λοιπόν θεσμικών εκτελεστικών οργάνων της Ένωσης. Η συζήτηση για την απαλλαγή δεν θα πρέπει κύριε Πρόεδρε να γίνει ένα πεδίο μάχης που ε, ανταλλάσσουμε επιθέσεις και πολιτικά σχόλια, ιδίως εν ώψη εκλογών. Νομίζω ότι στόχος της απαλλαγής είναι η τακτή και νόμιμη παλήθευση της εκτέλεσης ε, του προπολογισμού η εκτέλεση του προπολογισμού πρέπει να περιορίζεται σε αρχές της χρηστή μεσονομική διαχείρισης και αυτό είναι όλο. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό του Γενικού Γραμματέα τη Κομισιόν, κύριε Πρόεδρε. Ο Γενικός Γραμματέας τη Κομισιόν που υπενθυμίζω ορίστηκε το, Δεκέμβριο, το Φεβρουάριο του 2018, εγκρίναμε τον Απρίλιο ψήφισμα επ' αυτού και αυτή τη στιγμή παρόλα αυτά συζητάμε για την απαλλαγή του 17 δεν αντιστοιχούν όλα αυτά. Εγώ συμφωνώ με ορισμένου συναδέλφου, κύριε Πρόεδρε, ω προ το ότι το κοινοβούλιο είναι αυτό που θα πρέπει να εγκρίνει του λογαριασμού και την νομιμότητά του. Όμω, ε, απαιτείται μεγαλύτερη ηθική αξιοπιστία και νομιμοποίηση. Και αυτό θα το πετυχαίναμε εάν ε, είχαμε ε, δώσει το καλό παράδειγμα όλα τα θεσμικά όργανα με τον ορισμό των γενικών γραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ, και Κινίτσι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την εξαιρετική εργασία για την απαλλαγή του 2017. Θα ήθελα να αναφερθώ στους οργανισμούς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στον τομέα δικαιοσύνης, ε, μετανάστευσης, και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα διασυνοριακά εγκλήματα και αυτό μέσα στα πλαίσια και της αρχής της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής μέσα στα πλαίσια της διακυβέρνησης που εισαγάγει ο νέος ε, κανονισμός. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται διαφάνεια του προϋπολογισμού για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις έναντι των πολιτών. Ο κύριος Φίτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα μόνο ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Μετά από μία επιλογή πολύ συζητήσιμη και τη μεταφορά της έδρας στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, έχουμε τώρα ε, ένα κτίριο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο Άμστερνταμ και το οποίο είναι άδειο. Ενώ στο Μιλάνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα το κτίριο που ήταν διαθέσιμο. Όπως ξέρετε, στο Λονδίνο καταδικάστηκε ο οργανισμός σε, ένα, σε μια χρηματική ποινή αρκετά υψηλή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την επιλογή. Φαίνεται ότι είναι ένα ράπισμα προς τις επιλογές των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, Τζέλερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πρόεδρε, λένε... Ε, 60 χρόνια μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω ε, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης που συνδέεται και με τις ε, συμφωνίες ε, του Κοτονού που πάβουν να ισχύουν από του χρόνου ε, και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμη τι θα γίνει με το μέλλον αυτών των συμφωνιών. Πρέπει όμως να σκεφτούμε γενικώ το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχει άλλη θέση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και μέχρι στιγμής δεν είχαν καταφέρει να εφαρμοστούν πολλές φορές οι στόχοι αυτού του προγράμματος. Το διαπιστώ διαπιστώνει και το ελεγκτικό συνέδριο. Υπήρξαν παραλήψει, υπήρξαν προβλήματα και πολλές φορές είναι και πηγή ε, που τη χρησιμοποίησαν διάφορα καταπιστεύματα και νέα ταμεία και επομένω η διαφάνεια δεν υπηρετήθηκε ε, και η σωστή ε, εκτέλεση. Χαίρομαι με την πρόταση της Κομισιόν ε, μελλοντικά να περιληφθεί στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Αυτό είναι το θετικό γιατί έτσι θα υπάρχει και ο δέον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ευχαριστώ κύριο Σαντριέ για 1,5 λεπτό. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας θυμίσω την απόφαση Μάγερ. Διαβάζω άρθρο 11 του κανονισμού του προσωπικού που λέει ότι την εκτέλεση των καθηκόνων του ένας υπάλληλο δεν χειρίζεται υπόθεση στην οποία εμπλέκεται προσωπικός εμέσως ή αμέσω. Όμω, όπω όλοι γνωρίζουμε εδώ, ορισμός του κυρίου Σελμάγερ, ο Γενικού Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν αμφιλεγόμενη, τουλάχιστον. Και τα ερωτήματα είναι πολλά όσον αφορά τον διορισμό του. 24 Μαρτίου του 2018 συγκλήθηκε συσκέψη στο επιτελείο Juncker, στην οποία συμμετείχε ο κ. Σελμάγερ για το φάκελό του. Η απάντηση που δόθηκε δεν μας ικανοποίησε. Θέσαμε λοιπόν ερωτήματα, 61 τον αριθμό. Κατόπιν αυτών 2 Απριλίου του 2018, νέα σύσκεψη, επαναλαμβάνεται, στην οποία παρευρίσκεται και ο κ. Σελμάγερ για άλλη μια φορά. Πρέπει λοιπόν να το πάρουμε επίση, να το πάρουμε επιτέλου στα σοβαρά. Ο κ. Γιούνκερ δεν μα εξήγησε ενώπιον τη διάσκεψη των Προέδρων τι ακριβώ έγινε. Θεωρώ ότι πρέπει διαθεσμικά να δημιουργήσουμε μια επιτροπή έρευνα και εν μεταξύ προτείνω ο Γενικό Γραμματέα να παυθεί για να τηρηθούν όντω οι κανόνε που διέπουν τα θεσμικά μα όργανα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, έχουμε μόνο έναν ομιλητή στο πλαίσιο της διαδικασίας Κατστιάη. Δεν δώσω το λόγο σε άλλον. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι υπέρ της απαλλαγής και της έκθεσης. Θυμίζω ότι δυόμιση δισεκατομμύρια πήγαν σε κοινωνικέ επιχειρήσεις. Εδώ νομίζω μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Κυρίως με τη χρήση της πληροφορικής. Όμως, η προσθεμένη αξία των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι δεδομένη, είναι πασιφανής πλέον. Από εκεί πέρα να δούμε αν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Κάποιοι επικεντρώνονται στην Δημοκρατία τη Τσεχίας. Ε, δείτε όμως τι γίνεται και με του οργανισμού. Γιατί υπάρχουν διάφορα έργα οργανισμών όπου απασχολούνται άνθρωποι που έχουν συμφέροντα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν είναι διαφάνεια, αυτό είναι απαράδεκτο. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Έχουμε ψηφοφορία, ψηφοφορίε, μάλλον στι 5, οπότε πρέπει να κλείσουμε με τις παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό. Παρακαλώ. Ο κύριος Λέν, ο πρώτος ελεγκτικού συνεδρίου, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε και κύριοι βουλευτέ, καταρχά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και τι ε, πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσει. Σε δύο πτυχέ μόνο ε, θα αναφέρω. Η πρώτη αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και τα ευτικά ζητήματα. Θα ήθελα ε, να πω στην κυρία Μακοβέη ότι πράγματι υπάρχει αυτή η πρόθεση, το βλέπετε και στο έργο μα και όσοι ασχολείστε βλέπετε ότι η έκθεση για την κατάσταση των ηθικών κανόνων στα θεσμικά όταν θα είναι έτοιμη πριν από τις θερινές διακοπές και για μας ε, προβλέπεται έλεγχος μέσω ομοτήμων. Ένα peer review και ε, αυτό μάλλον θα είναι έτοιμο το peer review πριν το καλοκαίρι. Το δεύτερο θέμα Πολλές φορές ακούστηκε εδώ η επιθυμία ε, να, ε, σταματήσουν ε, τα σφάλματα, τα ποσοστά σφάλματος να μειωθούν. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι είναι ουσιαστικά, είναι στατιστική μαθηματική μέθοδος τα ποσοστά σφάλματος με κάποια βεβαιότητα, κάποιες πιθανότητες μπορούμε να υπολογίσουμε τι σφάλματα έχουν συμβεί και συνήθως ε, με βάση τα αποτελέσματα του σφάλματος που διαπιστώνουμε σε καμιά χιλιάδε ε, συναλλαγών κάνουμε αυτές ε, τους υπολογισμούς για το 2017 βασιστήκαμε σε αυτές τις αναλύσεις και είπαμε ότι είναι 2,4% το ποσοστό σφάλματος 95% πιθανότητες και συν πλήν 1% ανοχή διαφορά δηλαδή στην περίοδο τη 1,4 με 3,4 είναι αυτό το ποσοστό. Αν τώρα το σπάσουμε σε μικρότερα τμήματα, τότε θα έχουμε πολύ λιγότερα στοιχεία για να επεξεργαστούμε. Οπότε θα μειώνεται ακόμη περισσότερο ποσοστό σφάλματος. Δηλαδή αν έχουμε 0,9 ή 0,5 ποσοστό σφάλματος σε ένα διοικητικό τομέα. Αυτό είναι μια εκτίμηση. Ε, τίποτε περισσότερο ε, και μπορεί να αναφερθεί επί τα άνω, τα, ε, χείρο, επί τα αυτό το ποσοστό. Ε, επομένως ε, ε, είναι τόσο μεγάλη η γραφειοκρατική, διοικητική, το διοικητικό άχθο σε αυτό που δεν νομίζω ότι έχει το ε, νόημα που το, έχει κανένα νόημα. Ε, 45% ε, μπορούμε να καλύψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο ε, και βεβαίως ε, καταλαβαίνω ότι θέλετε ε, πιο ακριβή στοιχεία, πιο πολλούς κλάδους ε, και θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνω με αυτή την επιθυμία. Δεν γίνεται όμως γιατί επαναλαμβάνω αυτό είναι στατιστικό. Δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι περισσότερο. Δεν έχει κανένα νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Έτιγκερ έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, εγώ θα ήθελα ε, τρία βασικά πολιτικά ζητήματα να σχολιάσω εν συντομία εδώ. Το πρώτο άπτεται ενός συγκεκριμένου ε, ερωτήματος αν υπάρχουν ε, συγκρούσεις συμφερόντων ναι, και τι γίνεται με την τσεχική δημοκρατία. Από την αρχή Ιανουαρίου συγκροτήσαμε ομάδες εμπειρογνωμόνων για να δούμε τι γίνεται στη ΓΑΜΑ ΔΕΚΤΑ Ρέτζιο Άγκρι Employment και ε, υπάρχουν και άλλοι στην Πράγα ε, ε, ειδικοί οι οποίοι μελετούν όλο αυτό το φάκελο, τα στοιχεία, τα δεδομένα, όλες τις διαδικασίες και με αυτούς τους εμπειρογνώμονες τώρα προβαίνουμε στην αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων. Πρέπει να σας πω ότι παρακάλεσα τους συναντέλφους... και τους γενικούς διευθυντές των αρμοδίων αυτών υπηρεσιών πάρα πολύ γρήγορα αλλά και με πάρα πολύ μεγάλη ενδελέχεια να εργαστούν. Ε, δεν ε, μπορώ εγώ τώρα να σας πω όμως ε, ότι θα τους περιορίσω χρονικά γιατί θέλουμε να γίνει σωστή δουλειά και αυτό προηγείται, υπερτερεί του να βιαστούμε. Ε, πάντως ε, πιστεύω ότι σε λίγες εβδομάδες ε, θα και συγκεκριμένα στις 15 Απριλίου στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα παρουσιαστεί μια ενδιάμεση έκθεση πάρα πολύ αναλυτική για τους ελέγχους, τα audit και για τα πρώτα αυτά αποτελέσματα των εκτιμήσεων και εκεί μπορούμε να συναγάγουμε και κάποια αποτελέσματα. Παραλαμβάνω όμως χωρίς πίεση χρόνου γιατί θέλουμε να απαντήσουμε σωστά και ενδελεχώς σε όλα τα ερωτήματα. Δεύτερο σχόλιο σε ό,τι αφορά ε, το διαγωνισμό ή τέλος πάντων τον ορισμό ε, γενικού διευθυντού ε, πρέπει να σας πω ότι είμαστε πεπισμένοι ότι Υπάρχουν δύο δυνατότητες για την κατάληψη μιας θέσεως δηλαδή διαγωνισμός ή ο διορισμός και νομίζω ότι είναι εξίσου ε, και θα έλεγα και συμπληρωματικά ε, αποδεκτή αυτή, αυτές οι δύο δυνατότητες. Και υπάρχουν δύο πράγματα που είναι ενδιαφέροντα να απαφέσω. Πρώτα απ' όλα αυτές οι μεταφορές, τα transfers μπορεί να γίνουν πολλές φορές στην αρχή μιας θητείας, παραδείγματος χάρη ε, μιας νέας κομισιόν. Στην αρχή όμως μόνο, που μπορεί δηλαδή γενικούς διευθυντές να να τους ορίσει η Κομισιόν με αυτόν τον τρόπο. Με βάση βέβαια τις αρμοδιότητές τους και μπορεί να κάνει κάποιες ανακατατάξεις. Αυτό το λέμε transfer και είναι κάτι λογικό. Μπορεί να συμβεί και έναν κανόνα, ε, όχι όμως ε, μόνιμο και 100% έχουμε τον κανόνα της κινητικότητας κάθε 6-7 χρόνια υπάρχει αυτή η αλλαγή Τρανσφέρ και στην προκειμένη περίπτωση το λέμε. Και έχουν υπάρξει ε, τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα υπάρχουν κάποια παράπονα και καταγγελίες ε, όταν παραδείγματο χάρη 6, 7, 8 χρόνια ε, παρέμεινε στη θέση η ίδια Γενική Διευθύντρια για παράδειγμα και μου είπαν γιατί δεν την έχουμε αλλάξει. Ε, επομένως, ε, όλα αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες σε ό,τι αφορά τους ορισμούς, ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς να ε, γίνονται με τις σωστές διαδικασίες. Και το τρίτο θέμα το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι το αν και αν ναι γιατί σε ό,τι αφορά το Γενικό Γραμματέα. Ε, είχα πει το Μάρτιο στην Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού ότι υπάρχουν ε, πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. και ότι θα έπρεπε για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό να έχουμε λάβει ε, μέρος σε κάποιες από αυτές τις διαβουλεύσεις. Ε, και τις συζητήσεις. Από πότε ήξερε ο κ. Σελμάγερ ήταν μια ερώτηση. Από ποια ημερομηνία του ε, Φεβρουαρίου ήξερε. Αυτές τις ερωτήσεις ε, ο ίδιος μόνο μπορεί να τις απαντήσει. Εμείς δεν το ξέρουμε. Δυστυχώ, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι έναν όροφο πιο πάνω βέβαια ο Γενικός Γραμματέας ε, και μπορεί να ε, απαντήσει πάντως ε, ο ίδιος. Μόνο αυτός είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένη απάντηση σε πολλά από τα ερωτήματα τα οποία έθεσε το αξιότιμο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσάμπα έχει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για αυτή τη χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Χαίρομαι διότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζονται πολλές ανησυχίες καθώς και την ανάγκη βελτιώσεων για να υπάρχει ε, μία γνωμοδότηση, μία συνολική έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο που να συμπίπτει ως προς τα συμφέροντα όλων. Θα πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Παρά το γεγονός ε, του μηνύματος που αποστέλουμε στους πολίτες και τους φορολογούμενους, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αποδίδει τα αποτελέσματα, προσδοκόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν η κυρία Γιάλα Σέντερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ευχαριστώ για αυτή την τόσο εμπλουτισμένη συζήτηση. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Ε, νομίζω ότι δεν κατάλαβα τι εννοεί η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του προεπολογισμού σε σχέση με τις ΜΚΟ. Ξέρετε, κυρία Γκρέσλε, ότι εδώ μιλάμε και για τους πόλεμους στα Βαλκάνια όπου στη συνέχεια μετά τους βομβαρδισμούς έπρεπε να αποκατασταθούν οι υποδομές, ε, γέφυρες, ε, δρόμοι κλπ. Ε, δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη σύραξη των πόλεμων στα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι τα προβλήματα δεν άρχισαν το 2012 και δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έγινε με τις συμβάσεις που απορρίφθηκαν. Την κυρία Τάνια Γκρίνερ της ε, γνωρίζετε, την κυρία Τάνια Γκρίνερ τη γνωρίζετε πολύ καλά στο Σπίγκελ μίλησε ε, μακρόν για τις απαλλαγές και αυτό δείχνει τι πιστεύουμε ως προς τους πολίτες, ως προς το τη σύγκρουση συμφερόντων. Λυπάμαι κυρία Έτιγκερ, αλλά όταν ε, ο κανονισμός μας για την κατάσταση υπαλλήλων λέει στο, στο ότι ένας υπάλληλο στην άσκηση των καθηκόντων του δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με ζητήματα τη στιγμή που υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δρά αυτόνομα. Πρόκειται για το πρώτο τμήμα ενός μεγαλύτερου άρθρου. Ο κύριος Σέλμαϊερ ξέρουμε ότι έχει συγκεκριμένα συμφέροντα. Ευχαριστούμε ε, βάλει για δύο λεπτά. Διακόπτει ο πρόεδρος, την κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε στην, ε, από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θέλουμε να διαχειριστούμε καλύτερα εν γέννη τον προϋπολογισμό, αλλά γίνονται πολλές ε, άχρηστες δαπάνες ε, που αφορούν και τους ίδιους τους επιτρόπους, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις διοικητικές δαπάνες. Και κάτι άλλο για το επόμενο πι πι, επειδή υπάρχει μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης, ε, Γαλλία, Ιταλία, ε, Γερμανία ε, μέσα στα πλαίσια του ΟΑΕΠ θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έτσι ώστε οι επενδύσεις που φτάνουν σε προστιθέμενη αξία να μην υπολογίζονται, να μην συνυπολογίζονται στο έλλειμμα. Σμιτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα ολοκληρώνοντα τη συζήτηση. Θα ήθελα ο ρόλος επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να λαμβάνεται πιο σοβαρά υπόψη από ορισμένου συναδέλφου, διότι βλέπω ότι οι προτάσει και παρατηρήσει τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα εφαρμοστούν, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, αλλά αυτό ε, δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν για να κάνουν να, ε, να προβάλλονται κάποιοι συνάδελφοι ή για να ε, επιδιώκουν τους δικούς τους στόχους και να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για όλους και επομένως και τους συναδέλφους από όλους τους Ο κύριος Κόντε τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τις ηγητές για την πολύ καλή συνεργασία, αλλά να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες από τα άλλα θεσμικά όργανα, γιατί υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Όλους επίσης τους συνεργάτες και των γραμματείων θέλω να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Κύριο Σαρβαμά για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Η κατακλείδα. Πρόεδρε, συντομότατα γιατί ήδη προσέρχονται οι συνάδελφοι για τις ε, ψηφορίες και θέλω να δυσαρεστήσω κανέναν. Λοιπόν, αυτή η απαλλαγή είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν είναι ότι και ότι. Δεν αφορά τους οπαδούς του Brexit και τους ε, πολέμιους της Ευρώπης. Δεν είναι οι κραυγές περί πατάλης εδώ και εκεί. Το αντίθετο. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, στέλνουμε ένα μήνυμα. Ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε εδώ, ότι ελέγχουμε, ότι επιβλέπουμε, ότι επιτηρούμε το πώς δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτό το κάνουμε, πιστεύω, με επιτυχία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η κυρία Λαμπαγιώβα, δύο λεπτά, η τελευταία εισηγήτρια. Πρόεδρε, εγώ θέλω απλώ να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης για τη συνεισφορά τους και τη συμμετοχή τους στη σημερινή συζήτηση. Να παραλάβω ότι οι κοινωνικέ επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό το ρόλο στα κοινά και συμβάλλουν στην γνώση και την καινοτομία. Πρέπει να ενισχύσουμε επίσης τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προσφέρουν στην κοινωνία η καινοτομία δεν είναι προνόμιο μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων. Αντιθέτω και η ίδια έρευνα και ανάπτυξη θα ωφελήσει τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και τι κοινωνικέ επιχειρήσει. Θυμίζω την ομόφωνη υπερψήφιση των σχετικών στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολισμού. Πρόεδρο, πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε σήμερα στι 5, το οποίο σημαίνει σε 25 δευτερόλεπτα από τώρα. Ευχαριστώ.